την ε, έκθεση του κυρίου Τάκουλα σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών για τέσσερα λεπτά. Arvoisa puhemies, Euroopan unionin eettinen velvollisuus on... Σας ευχαριστώ πολύ. Η ηθική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μεριμνήσει ώστε όλα τα παιδιά, τα παιδιά επίσης παιδιά μεταναστών, να έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν μια καλή εκπαίδευση, καλή παιδεία. Κάθε παιδί πρέπει να έχει το δικαίωμα να έχει δωρεάν παιδεία εκπαίδευση, τουλάχιστον στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και χωρίς δαπάνες. Πρέπει να βελτιωθεί η γενική κουλτούρα του και να του δοθεί κάθε δυνατότητα να αναπτύξει τις ικανότητές του και να ενταχθεί στην κοινωνία και να μπορεί να υπομειστεί τις ευθύνες του ως ε, άτομο μέσα στην κοινωνία ώστε να είναι πλήρως πολίτης ε, με ε, όλα τα δικαιώματα στην κοινωνία αυτή. Έτσι λοιπόν οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει πάντα να λαμβάνουν υπόψη το καλύτερο δυνατόν για τα παιδιά. Η εκπαίδευση των παιδιών είναι σύνθετο έργο και των γονέων αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε είναι να πετύχουμε με τις προσπάθειες από κοινού όλων μας να βελτιώσουμε την προσωπικότητα και τις ικανότητες των παιδιών. Υπάρχουν πρόσφατες μελέτες για τα παιδιά μεταναστών που δείχνουν ότι συχνά η εκπαίδευσή τους ήταν αρκετά δύσκολη και αντιμετώπισε εμπόδια σε μια κοινωνία που σε σχέση με σχολεία βλέπουμε ότι ε, υπάρχουν σε πολλές τάξεις μόνο παιδιά μεταναστών. Με αυτόν τον τρόπο καταλήξαμε πολλές φορές οι οικογένειες να ε, φεύγουν, να παίρνουν το παιδί από το σχολείο της συνοικίας ώστε να καταλήγει σε ένα σχολείο παιδιών μεταναστών μεταναστών, αποκλειστικά παιδιών μεταναστών. Αυτό είναι κάτι το αξιολύπητο. Με αυτόν τον τρόπο το επίπεδο εκπαίδευση ε, και κατάρτιση των παιδιών είναι πάρα πολύ χαμηλό και ιδιαίτερα επειδή με αυτού του είδους ε, επικέντρωση σε ειδικά σχολεία για παιδιά μεταναστών αυτών των παιδιών δεν είναι καθόλου κατάλληλος ο τρόπος εκπαίδευσης ε, που τους παρέχεται και δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος για να ενταχθούν στις κοινωνίες μας, στα κοινωνικά μας συστήματα. Πρέπει να μεριμνήσουμε και να διασφαλίσουμε τα σχολεία να έχουν επαρκείς ε, πόρους, επαρκή κονδύλια αλλά επίσης και ποιότητα του εκπαιδευτικού δυναμικού, δηλαδή των δασκάλων και των καθηγητών και να μεριμνήσουμε επίσης να είναι επικαιροποιημένη η εκπαίδευση και η κατάρτιση που θα παρέχεται και ιδιαίτερα στην επόμενη φάση. Χρειαζόμαστε όχι μόνο αυτές τις προσπάθειες, ειδικέ προσπάθειες, αλλά και κονδύλια, επαρκή πρόσθετα, επιπρόσθετα κονδύλια για τα σχολεία και τους δασκάλους και καθηγητές. Και εδώ το θέμα της επικουρικότητας είναι δεδομένο. Τα κράτη-μέλη αποφασίζουν τι γίνεται. Αλλά επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του ανοιχτού συντονισμού έχει το καθήκον να ζητήσει να απευθύνει έκκληση στα κράτη-μέλη να δρουν με τον τρόπο που προπεριέγραψα. Διότι τα παιδιά των μεταναστών πρέπει να έχουν το δικαίωμα να μπορούν να έχουν την καλύτερη εκπαίδευση που θα τους προσφέρεται. Και έτσι θα μπορούν να εντάσσονται στα κοινωνικά συστήματα, στις κοινωνίες των χωρών υποδοχής. Γιατί διαφορετικά θα δούμε αυτό το οποίο συμβαίνει σε πολλές χώρες. Δεν θα ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους, θα έχουν ε, ε, δυσκολίες να ε, παρακολουθήσουν τις σχολικές τάξεις και έτσι θα περιθωριοποιούνται. Επιπλέον, Πρόεδρε, υπό το πρίσμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ε, ανθρώπων, των ατόμων, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά στα κράτη-μέλη τα οποία δεν επιθυμούν να πάνε σε άλλη χώρα να σπουδάσουν να, να, ή να εργαστούν επειδή γνωρίζουν ότι στις άλλες αυτές χώρες τα παιδιά τους δεν θα μπορούν να αποκτήσουν την αναγκαία παιδεία. Αυτό είναι απαράδεκτο όμω και δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε να συμβαίνει. Σε όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να παρέχεται επαρκέ επίπεδο εκπαιδευτικό στα παιδιά και ιδιαίτερα παιδιών, παιδιά μεταναστών. Πρέπει, αυτό είναι το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε και πρέπει σήμερα να μεριμνήσουμε να διασφαλιστούν οι όροι και προποθέσει τη εκπαίδευσή του και όχι να το αφήσουμε. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση που θα είναι η πιο κατάλληλη για το δυναμικό και τι ικανότητε. του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο στον, ε, ε, ε, στον Επίτροπο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να χαιρετήσω για αυτή την πρωτοβουλία και θα ήθελα κυρίως εξ ονόματος του συναδέλφου μου Γιάνν Φίγκερ να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Τάκουλα και την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε και το, κύριε και το γεγονός ότι στα κράτη-μέλη έχουμε παιδιά ε, μεταναστών που ε, έχουν ανάγκες να παρακολουθήσουν μαθήματα στα σχολεία είναι κύρια πρόκληση αυτή. Η εκπαίδευση είναι ουσιώδες στοιχείο για την ένταξη αυτών των παιδιών. Η απόκτηση γνώσεων είναι απαραίτητη διαδικασία όταν θέλουμε να διασφαλίσουμε διασφαλίσουμε την ένταξη αυτών των ατόμων σε μια κοινωνία. Μια κοινωνία που όλο και περισσότερο θα αντιμετωπίζει μια γενικότερη άμυλα και έναν γενικότερο ανταγωνισμό. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό το σχολείο να μπορεί έγκαιρα να διασφαλίζει τα θεμέλια τα εκπαιδευτικά ώστε να βελτιώνεται η συμβίωσή μας και να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα μεγάλα προβλήματα με, ε, για παιδιά μεταναστών στην Ευρώπη. Τα παιδιά μεταναστών αντιμετωπίζουν διπλή πρόκληση στην Ευρώπη σήμερα. Αφενός μη επαρκείς γλωσσικές γνώσεις ε, της γλώσσας πλευράς της χώρας υποδοχής, από την άλλη πλευρά δυσκολίες όσον αφορά τα σχολεία. Ε, πολλές φορές ε, σε σχέση με τα παιδιά γηγενών, τα παιδιά μεταναστών έχουν χαμηλότερους ε, βαθμούς και επιδόσεις στο σχολείο. Δεν μπορούν να ολοκληρώσουν την ε, εκπαίδευσή τους και έχουν και χαμηλότερο ποσοστό συμμετοχή σε αυτά τα μαθήματα. Τονίζεται από πλευρά τη εισήγηση πόσο είναι σημαντική η εκμάθηση τη γλώσσα τη χώρα υποδοχή, που πρέπει να υποστηρίζεται επαρκώ. Αλλά ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά πρέπει και η μητρική γλώσσα των μεταναστών αυτών, των παιδιών των μεταναστών αυτών να καλλιεργείται. Η συμμετοχή σε προσχολική εκπαίδευση και παιδεία είναι εξίσου σημαντική ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτά τα παιδιά στα συστήματα που έχουμε δημιουργήσει και έτσι να μειώσουμε τα κοινωνικά μειονεκτήματα τα οποία εφίστανται. Οι δάσκαλοι θα πρέπει να έχουν τις αναγκαίες, τα αναγκαία προσόντα ώστε να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα της πολυπολιτισμικής προσέγγισης. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει και ένα σημαντικό στοιχείο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και κατάρτισης των δασκάλων και καθηγητών. Χαίρομαι για το σε αυτό το σημαντικότατο θέμα υπάρχει σύμπτωση απόψεων και συνένεση. Τώρα σημαντικό είναι αυτές οι καλές προθέσεις χειροπιαστά να πάρουν σάρκα και οστά, ώστε πραγματικά να βελτιώσουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για τα παιδιά μεταναστών. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη για να αναβαθμιστεί η ποιότητα που παρέχεται στην εκπαίδευση για αυτά τα παιδιά και ταυτόχρονα δραστήρια να συμμετάσχουμε ώστε να προωθηθεί η κοινωνική ένταξη αυτών των παιδιών. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη ώστε να είναι δυνατόν στα σχολεία να αντιμετωπιστούν αυτές οι πολλαπλές προκλήσεις ώστε να είμαστε σε θέση της προκλήσεις της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικής κοινωνίας ε, να τις εκμεταλλευτούμε μέσα από τα σχολεία αυτά ε, προς όφελος των παιδιών. Φυσικά το περιεχόμενο των μαθημάτων και τα σχολικά φορολογικά συστήματα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν έχει πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με οποιονδήποτε τρόπο να αναμειχθεί σε αυτά. Όμως θέλω επίσης να πω ότι η επιτυχής ένταξη των παιδιών μεταναστών την Ευρώπη συνολικά την αφορά στο σύνολό της Έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά ο ένας, από τον ένα, ο ένας από τον άλλο και μπορούμε να μάθουμε πολλά ο ένας από τον άλλο και είμαστε βέβαιοι ότι η έκθεσή σας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για να καταδειχθεί τι πραγματικά συγκεκριμένα μπορεί χειροπιαστά να γίνει ώστε τα κράτη-μέλη να υποστηριχθούν σε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ. Merci Ευχαριστώ. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Τώρα έχουμε μία σύντομη παρουσίαση της έκθεσης Βαλέαν για την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των Ευρωπαίων πολιτών και των οικογενειών τους στην επικράτεια των κρατών μελών.